Uh, Καλημέρα σε όλους. Έχει περάσει ένα τέταρτο. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έγκριση της μερίσιας διάταξης. Υπάρχουν ενστάσεις. Θα κάνουμε μια αλλαγή στο σημείο 4 για την πρόεδρο των τριμερών διαπραγματεύσεων η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα μετά από το σημείο 19 και μία-δύο ψηφοφορίες θα προσθεθούν κατά πάσα πιθανότητα στην ώρα των ψηφοφοριών ε, ανάλογα με αποτέλεσμα των ε, τριμερών συνεδριώσεων για το GSPM και τα EITs. Πρακτικά τώρα της τελευταίας ε, συνεδρίασης, ο συνήθως θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται εκτός και αν υπάρξουν σχόλια πριν από το πέρας της ε, συνεδρίασης. Και πάμε τώρα στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο συνήθως. Και σας έχουν διανεμηθεί και τα θέματα της ε, συνεδρίασης και της αλληλογραφίας. Για το σημείο 4 είπαμε η πρόεδρος των τριμερών διαπραγματεύσεων. Το περάσαμε προηγουμένως ε, όπως σας είπα στο σημείο 19 και πάμε στο σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων με τον Μάικολ Γκούσταυσον, ο οποίος κάθεται εδώ ξεφωνήμων και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών και θα συζητήσουμε μαζί του τα θέματα ενσωμάτωσης τη διάθεση του φίλου στι εργασίε των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Σα καλωσορίζουμε. Όπω γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξορθολογιστούν αυτές οι προσπάθειες ε, στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο προσκεκλημένος μας σήμερα, όπως σας είπα, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών. Θα του δώσω λοιπόν απευθείας το λόγο προκειμένου να μας πει τις απόψεις του για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στη συνεδρίασή σας. Θα περάσω στα σουηδικά, διότι είναι λίγο πιο εύκολο για μένα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Φορέστε τα ακουστικά σας λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση λοιπόν στην συνεδρία της Επιτροπής σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ και μπορώ να σας πω πώς εξελίσσονται οι εργασίες μας, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τη διάσταση του φύλου σε όλα τα θέματα τα οποία μας αφορούν. Στην Επιτροπή Γυναικών έχουμε μια διτή προσέγγιση ένα διτό τρόπο αντιμετώπισης ε, των θεμάτων ε, που αφορούν ε, την ισότητα. Αφενός μας ενδιαφέρει το να επισημάνουμε τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να βρίσκεται αυτό στην προτεραιότητα της, του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε συνεχώς να ενσωματώσουμε τη διάσταση του φίλου σε όλες ε, τις πολιτικές ε, ε, τοποθετήσεις μας. Αυτό το οποίο αποκαλούμε gender mainstreaming. Βάσει τη συνθηκή της Λισαβόνας, στο άρθρο 8 αναφέρεται η αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να άρει οποιαδήποτε ανισότητα υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή είναι η νομική μας βάση. Γι' αυτό ε, και εδώ ε, και στη δική σας την Επιτροπή παρουσιάζουμε τροπολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους το θέμα της ισότητας των φύλων. Υπάρχει ένα δίκτυο εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο φροντίζει να υπάρχει ένα μέλος σε κάθε ε, επιτροπή το οποίο είναι επιφορτισμένο να διασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο, διότι κάποιοι δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς μπορεί να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου σε όλα τα θέματα, αλλά με πείρα και με ε, ε, συνεχή προσπάθεια μπορούμε να εντάξουμε αυτή τη διάσταση του φύλου σε όλες μας τις πολιτικές. Πέραν αυτού, κάθε δεύτερο χρόνο γίνεται μία έρευνα η οποία αποστέλλεται σε όλες τις επιτροπές ε, για να δούμε ε, αν λειτουργεί αυτή η πολιτική. Βλέπουμε τι στρατηγικές έχουν εφαρμοστεί και κατόπιν όλα αυτά μαζί τα εξετάζουμε και εξακολουθούμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που διαπιστώνονται σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου. Ε, Έχουμε και ένα σχετικό ψήφισμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς ασχολούνται ε, οι διάφορες επιτροπές με τα θέματα του φύλου και πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Με χαροποιεί λοιπόν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Επιτροπή σας ε, ε, επέλεξε τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ως υπεύθυνο για τα θέματα αυτά, διότι είναι σημαντικό αυτό το καθήκον και δείχνει πόση σημασία δίνετε εσείς στο θέμα αυτό. Είναι επίση πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να αποτελούμε πρότυπο για όλες αυτές τις πολιτικές. Θα πρέπει να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταθούμε στο ύψο των εργασιών μας, διότι υπάρχει σχετικό στόχος και στη συνθήκη τη Λισαβόνα και δηλώνεται ρητός. Θεωρώ λοιπόν ότι αποτελεί πάρα πολύ καλή βάση για να βλέπουμε τα θέματα τη ισότητα, αλλά και πέραν αυτού στην πράξη θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε πολύ σκληρά να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνεται πάντα υπόψη η διάσταση του φύλου σε οτιδήποτε κάνουμε. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή σας προκειμένου να προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Εγώ έχω προωθήσει τέσσερις βασικές ιδέες. Καταρχάς, κάθε Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει μια στρατηγική για το φύλλο, προκειμένου να καθορίσει επακριβώς πόσο σημαντικές θα είναι αυτές οι σχέσεις ε, ε, και πώς συνδυάζονται με τα θέματα τα οποία συζητάτε. Κατόπιν, θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσεις πρωτοβουλίες που επισημαίνουν τις ε, προοπτικές ε, του φύλου. Παραδείγματος χάρη, γυναίκες στο διεθνές εμπόριο. Μια τρίτη δυνατότητα είναι ότι θα πρέπει να προσπαθείτε συνεχώς να ενισχύσετε τη συνεργασία με τις υπόλοιπες επιτροπές ώστε να υπάρχουν συμπληρωματικά ε, στοιχεία ε, για κάθε επιτροπή σε θέματα φύλου. Και το τέταρτο στοιχείο είναι να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει εδώ στο Κοινοβούλιο και να εφαρμόζονται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι και χαίρομαι που επιλέξατε και μένα και με καλέσατε εδώ για να σας ε, πω τη δική μου εμπειρία και την να, σας, να μοιραστώ μαζί μου την εμπειρογνωμοσύνη σας. Υπήρχε ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε τον Νοέμβριο για την ενίσχυση της διάσταση του φύλου σε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του ψηφίσματος θα πρέπει να κάνουμε μία απόπειρα να αλλάξουν οι δομές μας ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η διάσταση του φύλου είναι πανταχού παρούσα στις εργασίες μας. Στο ψήφισμα αυτό αναφέρεται ότι η αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Γυναικών είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να καταθέτει τροπολογίες στις ε, υπόλοιπες επιτροπές. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο να σας πω ότι εμείς με τα χαράς να καταθέτουμε σχετικές τροπολογίες για τα θέματα του φύλου, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ε, να το υλοποιήσουμε χωρίς να πρέπει κάθε φορά να είμαστε εμείς αυτοί που σας πιέζουμε. Προσβλέπω λοιπόν ε, στην ημέρα που η κάθε επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τη τη διάσταση του φίλου μόνη τη και δεν θα πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα σας πιέζουμε κάθε φορά. Αυτά λοιπόν προς το παρόν και είμαι στη διάθεσή σας για ιδέες και προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας και μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσει τώρα. Να σα πω Δευτή επιτροπή έχει 31 πλήρη μέλη. Μόνο 7 όμως είναι εδώ. Οι υπόλοιποι λείπουν. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματική εικόνα της Επιτροπής μας. Και Συμμετέχουν πολλοί οι γυναίκες ε, και στις, ε, στην εκπόνηση εκθέσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό σύμφωνο με την ε, πολιτική περί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω μαζί μου τα συγκεκριμένα στοιχεία. Any question, any remark, any... Ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Ο κύριος Σόλτς. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας και φαντάζομαι είναι πολύ σημαντικό θέμα εφόσον έχει γίνει λόγος για την οριζόντια γραμμή και το mainstreaming. Συχνά το συζητάμε αυτό ε, καθώς και το θέμα των γενών, αλλά αν ε, μιλά κανείς και για οικολογικά θέματα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο mainstreaming. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία μέσω της οποίας συνδέονται διάφορες πολιτικές. Συχνά έχουμε βέβαια να κάνουμε με μια κατάσταση όπου κρίνουμε από τις εξελίξεις ε, στον επιχειρηματικό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα του εμπορίου, στην... επίπτωση μάλλον του εμπορίου απευθείας στις γυναίκες. Αφού είδαμε τη διαδικασία στην Επιτροπή Γυναικών σε σχέση με τις τροπολογίες περί gender mainstreaming στις υπόλοιπες εκθέσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας, οι εμπειρίες σας σε σχέση με την πραγματικότητα σε άλλες επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα. Εσείς μόλις εξηγήσατε τη γενική σας προσέγγιση, αλλά ποια είναι η εμπειρία σας, γιατί για να είμαι ειλικρινής, συχνά στις εκθέσεις μας δεν είναι το θέμα του gender mainstreaming τη βασική μας ε, ανησυχία. Βέβαια σκεφτόμαστε αν θα έχει αντίκτυπο στην ισότητα των φίλων, στα παιδιά και τα λοιπά η κάθε οδηγία μας, αλλά πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ξέρουμε τι αναμένεται από την Επιτροπή μας σε σχέση με τις προκλήσεις που σας απασχολούν. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση. Πριν να δώσω πάλι το λόγο στον προσκεκλημένο μας, θα ήθελα να σας πω ότι ανταποκριθήκαμε στο εκδαμένο ερωτηματολόγιο που προετοίμασε η Επιτροπή των Γυναικών και η Αντιπρόεδρος μας Χριστιάνα Μουσκαρδίνη είναι υπεύθυνη για αυτήν την διάσταση της εργασίας μας στην Επιτροπή και τη συνεργασία μαζί σας δηλαδή. Κύριε Γκούσταυσον, έχετε πάλι το λόγο. Eh, eh, σας ευχαριστώ. Όντως, αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας ποια είναι η δική μας ευθύνη όσον αφορά την υποβολή αυτών των τροπολογιών και τις δικές μας συμβολές. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι πολύ ικανοποιητική η κατάσταση. Όταν εμείς ως Επιτροπή διαβάζουμε τις προτάσεις που προέρχονται από τη δική σας Επιτροπή ή από άλλες, έχουμε την αρμοδιότητα να πούμε ναι, εδώ λείπει μια προοπτική περί φύλων, αλλά δεν έχουμε τις ε, απαραίτητε γνώσεις ας πούμε, του δικού σας πεδίου του διεθνούς εμπορίου. Όταν μιλάμε λοιπόν ε, για τις ε, απαιτήσει μας όλα γίνονται υπό το φως των δικών μας αρμοδιοτήτων και όταν κανείς δει τη δική μας συμβολή ίσως και να σκεφτεί όταν εσείς ας πούμε, το βλέπετε ναι μα Εντάξει, ε, ναι, συμφωνούμε αλλά, επί της αρχής, αλλά η διατύπωση είναι πολύ παράξενη. Άρα το καλύτερο θα ήταν η δική σας επιτροπή να δεχτεί εξ αρχής μια προοπτική περί φύλων. Γιατί εσείς γνωρίζετε το θέμα σας. Εμείς ε, αντίθετα γνωρίζουμε τη διάσταση της ισότητας. Αν όμως εξ αρχής μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά ήδη στο κείμενό σας, τότε εντάξει, θα ήταν πιο καλά. Δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο ε, σαν να προσπαθούμε να βάλουμε μια ε, σφίνα περί φύλων, το οποίο όμως δεν είναι το καλύτερο, γιατί εσείς γνωρίζετε τα θέματά σας και εσείς μπορείτε να ξέρετε καλύτερα ποια μπορεί να είναι η προοπτική του φίλου μέσα στο πλαίσιο και της ισότητας στις δικές σας εργασίες. Γιατί πολλές φορές ε, ε, σκεφτόμαστε ναι, αλλά αυτό το, έχουμε, το έχουν σκεφτεί οι γυναίκες. Μα το θέμα της ισότητας δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αυτό το θέμα είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Και φυσικά αφορά και τις γυναίκες και τους άνδρες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως δεν πρόκειται για μια προοπτική ε, που αφορά ένα κομμάτι. Αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θα ήταν καλό λοιπόν να μην χρειάζεται καν η Επιτροπή μας να γράφει αυτές τις τροπολογίες για το gender mainstreaming, αλλά να το έχετε αυτό υπόψη σας εξ αρχής. Συμφωνώ βέβαια ότι δεν είναι προφανέ κάτι τέτοιο. Εγώ έχω δουλέψει για αυτά τα θέματα εδώ και 20 χρόνια. Αλλά πριν να φτάσω σε μια προπτική του gender mainstreaming για όλα τα θέματα και εγώ ίδιο χρειάζεται να το σκεφτώ ε, επί μακρόν. Και μα, έμαθα σιγά σιγά πώ γίνονται όλα αυτά. Αλλά αν μπορέσετε να εισάγετε αυτή τη στρατηγική στη δουλειά σα, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο απλά όλα και δεν θα χρειαζόταν να ασχολείστε με, τα δικά μας, ε, με τις δικές μας τροπολογίες. Και επειδή για ακόμη μια φορά λέω δεν έχουμε τις συγκεκριμένες γνώσεις που έχετε εσείς για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κουσαυσόν για την σημερινή του παρουσία εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα που δεν συνδέεται άμεσα με το διεθνές εμπόριο. Ε, το ερώτημά μου λοιπόν δεν άπτεται άμεσα του διεθνούς εμπορίου, αλλά θέλω να πω ότι διαπιστώνω με χαρά ότι και εσείς αναγνωρίζετε τη σκληρή δουλειά που κάνουμε στην Επιτροπή μας για αυτά τα ζητήματα που θέσατε. Ένα θέμα που ίσω παραγνωρίζετε καμιά φορά είναι ότι μένουν και οι άντρε στο περιθώριο. Δεν θέλω τώρα να βγω εκτός θέματος, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί και εσά, δηλαδή ότι μια φορά παραγνωρίζει το ρόλο των ανδρών. Βλέπετε κάποια στοιχεία, για παράδειγμα, και πώς επηρεάζει α, αυτό το φαινόμενο το εμπόριο. Για παράδειγμα, ζούμε από την προώρια εγκατάλειψη του σχολείου α, σε αγόρια και κορίτσια. Αν δείτε πόσα κορίτσια, το ποσοστό των κοριτσιών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια α, εκπαίδευση, θα δείτε ότι υπάρχει μια δυσαναλογία ανάμεσα στον υψηλό αριθμό των κοριτσιών και το πολύ χαμηλότερο α, των αγοριών. Αυτό είναι κάτι που σε έχει απασχολήσει ως ε, παράγοντας που επηρεάζει το εμπόριο μεταγενέστερα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ο παράγοντας συνιστός άνδρας. Παραγνωρίστε αυτές τις παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, θα θέλετε να απαντήσετε, κύριε Γούστευσον. Ναι. Βεβαίως. Να επαναλάβω πρώτα απ' όλα αυτό που είπα και νωρίτερα. Όταν μιλάμε για θέματα ποιότητας, δεν περιοριζόμαστε βεβαίως και μόνο στις γυναίκες. Θέλουμε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους, για άνδρες και γυναίκες, ε, να έχουν ε, τη δυνατότητα να ασκήσουν όλοι το δικαίωμά τους ε, στη συμμετοχική δημοκρατία. Έχετε δίκιο, λοιπόν, η πρόορια κατάληψη του σχολείου και η αποτυχία, αν θέλετε, ε, στο σχολείο που αφορά κυρίως ε, τα αγόρια είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Και στη δική μου χώρα τα αγόρια καταγράφουν λιγότερο καλά, αν θέλετε, αποτελέσματα και επιδόσεις στο σχολείο σε σχέση με τα κορίτσια. Όταν μιλάμε για ανισότητες, ε, δεν, μιλ... δεν μόνο στις γυναίκες. Εννοείται ότι πρέπει να δούμε το θέμα σφαιρικά. Παρά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όταν μιλάμε για ανισότητες, κατά κύριο λόγο το φαινόμενο α, και πλήττει τις γυναίκες. Είναι ένα γεγονός και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή υπάρχει ακόμη μεγάλος δρόμος ε, μπροστά μας για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για άσκηση των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών αλλά και ισότητας των Φίλων. Το λέω και το επισημαίνω και ισότητα των Φίλων. Well, the name of the committee is still It means... Ναι, αλλά η Επιτροπή φέρει πρώτα απ' όλο τον τίτλο ε, Επιτροπή Γυναικών, έτσι δεν είναι, εκεί δίνεται το ιδιαίτερο βάρος. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε τα πέντε θεματάκια σήμερα και αύριο να ε, επεξεργαστούμε. Λοιπόν, το σημείο 6. Εδώ έχουμε να κάνουμε τροποποίηση τριών κανονισμών που αφορούν την εισαγωγή ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία. Όσον αφορά την ευθυγράμμιση των κανονισμών αυτών με την διαδικασία επιτροπολογίας. Είμαι εγώ ίδιος ο εισηγητής. Θα ήθελα εντάχει να σας ενημερώσω τι έκανα σε αυτό το σχέδιο κειμένου να σας παρουσιάσω λιγάκι τη φιλοσοφία πάνω στην οποία εδράζεται το κείμενό μου. Αφορούν το Omnibus 1, νομοθεσία σε σχέση με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και Omnibus 2. Έχετε ενώπιόν σας ε, το σχέδιο έκθεσης. Παρακαλώ τα σχόλιά σας, ε, παρατηρήσεις ή ενστάσεις. You might be willing to Θέλετε παρακαλώ να σχολιάσετε. I have not yet... Uh, δεν ε, έχω υποδείξει. Όχι, έχω μίλησα με τους κοιόδης, αλλά δεν είναι κανόνας από τους κοιόδης συζητητέ εδώ. Μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να σχολιάσει. Listen to the commission. Να ακούσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κυρία Ντάρμαλ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, I'll be very brief. Θα είμαι συνοπτικότατη. Η Κομισιόν διαφωνεί για τις τραυπολογίες 1, 3 και 7 διότι δεν συνάδουν με την ε, συνεννόηση στην οποία είχαμε καταλήξει. Ειδικά όσον αφορά τις 1 και 3 υπάρχει μια αιτιολογική σκέψη ε, το σημείο 4 της κοινή συνεννόησης ε, και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να παραμείνει και να μην αλλάξει. Για την τροπολογία 7 τώρα θα θέλαμε να εφαρμοστεί ο καταρχήν χρόνων για τις εστάσεις που είναι δύο μήνες και όχι τέσσερις μήνες. Κατά τα άλλα συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σημειώνουμε τις διαφωνίες σας. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 1η Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Και εγώ θα λάβω υπόψη μου και τις ενστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν υπάρχει κάποια διαφορά θα καταθέσω τροπολογίες στο σχέδιο εκθεσής μου. Να περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7. Και πάλι νομοθετικός φάκελος, τροποποίηση του κανονισμού του 1994 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόλιο κρέα υψηλή ποιότητα το χείριο κρέα, το κρέα πουλωρικών, το σιρτάρι και το σιμιγδάλι, καθώς και τα πίτουρα και βγαίνει άλλα υπολείμματα. Έχετε και πάλι το σχέδιο έκθεσης, ο υποφαινόμενος είναι ο εισηγητής. offer the merits of my draft report. Uh, Δεν έχω τίποτα να αλλάξει στο σχέδιο έκθεσή μου. Να δώσω το λόγο στα μέλη τη Επιτροπή για να σχολιάσουν. Ε. Δεν βλέπω κάποιον να θέλει να σχολιάσει. Οι σκιώδη συζητητέ και πάλι απουσιάζουν. Ο λόγος και πάλι στην Επιτροπή λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για την έκθεσή σας για τους ίδιους λόγους που μόλις σας εξέθεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί τις τροπολογίες 1 και 5 Ευχαριστώ Χωρίς μικρόφωνο Στο σημείο 8 τώρα, ο εισηγητής απουσιάζει, ο κύριος Πιέλνερ. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 9. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κυργυσίας. Και πάλι εγώ είμαι ο εισηγητής νομοθετικός φάκελος και πάλι. Έχετε το σχέδιο έκθεσης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα ε, γράφονται στην έκθεση. Το βασικό ζήτημα είναι πολιτικής φύσεως και είναι και πάλι το θέμα της επιτροπολογίας φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ε, πει τις ενστάσεις της. Πριν δώσω το λόγο όμως στην Επιτροπή, να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Σχόλια. Όχι. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο κύριος Τέξ, άρτη αφιχθής. Ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο, το θέμα ήταν να συζητηθεί λίγο αργότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Όλα φαίνεται οφείλονται στο πόσο αποτελεσματικός είστε η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική λόγω της πολιτικής κρίσης που έπληξε τη Δημοκρατία της Κυργισίας το 2010 και τα επεισόδια τα οποία είχαμε στη συνέχεια. Σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση, η χώρα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα παρά τις προκλήσεις, ε, κατάφερε να μπει στο δρόμο της δημοκρατικής μεταρρύθμισης, ενεκρίθη ένα νέο σύνταγμα, έγιναν και νέες κοινοβουλευτικέ εκλογές και προεδρικές εκλογές πέρσι. Και για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας, ώστε να βοηθήσουμε τις αρχές οι οποίες είναι υπέρ της δημοκρατίας να προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Έγινε μια διάσκεψη χορηγών το 2010 και λήφθηκαν και αιτήματα για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησε σε ένα πρόγραμμα με τη χώρα και γι' αυτό και εμείς μετά από αυτό προτείναμε αυτή τη μακροοικονομική συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία ε, προτείνουμε να δοθούν κατά το ίμιση μέσω επιδοτήσεων. Εσείς κύριε Πρόεδρε ζητάτε να διαγραφεί η χρήση της συμβουλευτικής διαδικασίας ε, στην αιτιολογική σκέψη 13 που δεν δημιουργεί μεν πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία. Το βασικό όμως για μας είναι ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει μια συμβουλευτική διαδικασία ε, ή μια συνήθις διαδικασία και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί για τα μνημόνια συνεννόησης. Προς το παρόν λοιπόν ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, οποιαδήποτε από αυτές τις προτάσεις, δεν μπορεί να εγκριθεί καμία πρόταση και όπως γνωρίζετε αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και για την πρόταση για τη Γεωργία. Εκεί έγινε πρόταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ιανουάριο του 2011 και δεν έχει ακόμα επιληθεί το θέμα της επιτροπολογίας. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να, βρεθούμε μια, να βρεθεί μια λύση σε αυτή τη διαδικασία για να μην σταματήσουν και οι υπόλοιπε ε, προτάσεις μακροοικονομικής χρηματοδότησης χρηματοδοτική συνδρομής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και λόγω του περιβάλλοντος που ζούμε αυτή τη στιγμή και για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που είχε η Αραβική Άνοιξη στην ε, ε, προς νότο γείτονα περιοχή. Παραδείγματο χάρη, η Αίγυπτο ζήτησε χρηματοοικονομική συνδρομή τη τάξη των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ετοιμάζουμε την πρόταση σε συνεργασία με τι Αιγυπτιακέ Αρχέ και ελπίζουμε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την πρόταση αυτή μόλι υπάρξει πρόγραμμα από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και έχει συμφωνηθεί. Και από εκεί αναμένονται και πάλι κάποιε καθυστερήσει λόγω τη πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο. Για να επανέλθω τώρα στην Κυργυσία. Ελπίζουμε να είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε με το Συμβούλιο για το κατά πόσο θα υπάρξει μια συμβουλευτική διαδικασία ή μια διαδικασία εξέτασης. Ε, για μας ε, το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε είτε να συζητηθεί στο πλαίσιο αυτής της πρότασης για την Κυργησία ή στο πλαίσιο της πρότασης για τη Γεωργία, αλλά οποιαδήποτε λύση ούτως ή άλλως θα είναι ενδιάμεση μέχρι να υπάρξει μια συνολική συμφωνία ε, στα πλαίσια του βασικού κανονισμού και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πολύ γρήγορα ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτή η χρηματοοικονομική συνδρομή για να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες οι οποίες είναι και στενά συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Συμφωνούμε ότι είναι η επίτευξη συμφωνία σε αυτό το θέμα επίγουσες ανάγκης. Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για το πολύ περίπλοκο θέμα της επιτροπολογίας. Να σας θυμίσω το πλαίσιο, ε, όπου ο εισηγητής, ο κύριος Κάζακ, έχει προτείνει αντί τις εφαρμοστικές πράξεις να έχουμε κατεξοδότηση πράξεις για τη συνειοθέτηση του Μνημονίου Συνεννόησης. Δεν είναι εύκολο λοιπόν το θέμα. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 1η Ιουνίου το μεσημέρι στις 12. come back to Helen's report item 8 because he is not still there. So what should we do? Ε, για το σημείο 8 δεν μπορούμε να επανέλθουμε γιατί ο εισηγητής δεν έχει φτάσει ακόμα. Σε. Να περάσουμε στο σημείο 10 τότε. Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας και του Περού. Διαδικασία συνένεσης. Ο συγητής μας είναι ο Μάριο Ντάβιντ από το ΕΛΚΑ και το σχέδιο σύστασής του είναι στα σφακέλους σας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή τον Μάριο Ντάβιντ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος γιατί έχουμε ήδη συζητήσει ε, το θέμα και θα το ψηφίσουμε το απόγευμα ένα ψήφισμα, ένα ενδιάμεσο ψήφισμα για το θέμα αυτό και γι' αυτό νομίζω πως έχουμε καλύψει πάνω κάτω τα θέματα που μας ανησυχούν και τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το στάδιο. Να σας θυμίσω το γεγονός ότι επισήμως, αν και πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων περί συνένεσης, το θέμα είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα ε, κληθεί από το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Ε, από ό,τι ξέρω ακόμα συνεχίζονται οι υπογραφές αυτό το μήνα. Περιμένουμε λοιπόν από το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την εργασία του, όπω ίσω φαντάζεστε μετά από την ψηφοφορία που θα γίνει απόψε και από τον Ιούνιο στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, θα... Επειδή δείξαμε την ανησυχία μας σε σχέση με την παρακολούθηση τη συμφωνία αυτή ε, από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει, για δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα και ε, τις ε, συναλλαγές τα οποία εξηγώ και στην επεξηγηματική μου σημείωση δεν θα σας εντυπωσιάσει ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα ζητήσω από το Κοινοβούλιο να δώσει τη συνένεσή του για αυτή την εμπορική συμφωνία. Όπως ξέρετε ο κ. Ζολάνγκη και εγώ ως εισηγητής ε, εισηγητές των δύο εκθέσεων σε σχέση με αυτό το θέμα, τη συνένεση και την ρήτρα ασφαλεία, θα τα εκφεύγουμε αύριο για την Κολομβία και το Περού. Και αν συμφωνείτε και αν ε, συμφωνεί και ο κύριος Λάγκη βεβαίως, θα σας φτιάξουμε έκθεση που θα σας υποβάλουμε αν θέλετε βέβαια να τη βάλετε στην ατζέντα της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Ντάβιντ... Έχουμε το πακέτο το συνοδευτικό για την Κολομβία και το Περού και εδώ χρειάζεται να γίνουν κάποιες ε, διευκρινήσεις. Η συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο ίσως να είναι ε, πιο ε, σκληρή σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Ξέρουμε ποιες θα είναι οι θετικές πτυχές μιας εμπορικής συμφωνίας με το με την Κολομβία και το Περού, ωστόσο τα πλονεκτήματα και τα ωφελήματα θα πρέπει να φτάσουν και στους πληθυσμούς των χωρών αυτών και γι' αυτό θα θέλαμε παράλληλα να αναπτύξουμε έναν οδικό χάρτη με τα κοινοβούλια της Κολομβίας και του Περού, ακριβώς έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και να καλυφθεί και αυτή η ανησυχία μας. Αυτή είναι μια προϋπόθεση για να έχουμε μια, να δώσουμε μάλλον τη συνένεσή μας σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Χαίρομαι λοιπόν για τη συμφωνία για αυτήν τη διαδικασία. Θα συζητήσουμε με τους εταίρους, με τις κυβερνήσεις, ε, τα κοινοβούλια της Κολομβίας και του Πέρου για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση. Και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης και των διαπραγματεύσεων που θα κάνει ο, ο Ντάβιντ. Θα μιλήσουμε και για τον κανονισμό ασφαλείας και θα συζητήσουμε εις βάθος για την εμπορική συμφωνία. Για την αξιολογήσουμε. Ε, είμαι, λοιπόν ικανοποιημένος που υπάρχει συμφωνία για αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ο Σόλτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές για την ε, ήδη μακρά τους, ανά του μήνα νομίζω, συνεργασία. Έχουμε ανταλλάξει ε, πολλές φορές απόψεις όσον αφορά αυτή την ε, συμφωνία ή μάλλον τον, το εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας συνεργασίας. Και νομίζω πως ήδη έχουμε μπει στον έλεγχο αυτής της συμφωνίας Μα θυμήσατε πως επισήμως δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει τις συζητήσεις γιατί αυτή η συμφωνία θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Αμερική και όλα αυτά τα θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις γενικότερες πτυχές αυτής της συμφωνίας να πω ότι Ήδη έχει γίνει συμφωνία, ε, μάλλον ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τι οικολογικέ τυχέ, τον αντίκτυπο στου ε, γηγενεί, και θέλω να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Πρεσβείας που έχει επίσης ε, συνοδέψει τις ανταλλαγές απόψεων στην Επιτροπή σε σχέση με αυτές τις διάφορες πτυχε. Και πάλι ωστόσο θα ήθελα να <clears throat> αναφερθώ σε τρία σημεία τα οποία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ακροάσεων που είχαμε ακούσαμε πολλούς εκπροσώπους να μιλούν για τις, ε, τον αντίκτυπο της εμπορικής συμφωνίας για τους στοχότερους και για το περιβάλλον στις δύο αυτές χώρες και ε, Κολομβία και Περού και πιο συγκεκριμένα με τις στρατηγικές των εξορυκτικών βιομηχανιών που όπως είδαμε ως αποτέλεσμα της ε, μελέτης ε, αντικτύπου, θεωρούμε πως η εμπορική αυτή συμφωνία θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις ε, για τους φτωχούς και για την οικολογία. Να πω επίσης ότι η εκτός από την εξωτερική βιομηχανία αλλά και οι καλλιέργειες ε, γεωργικών καυσίμων ε, είναι πολύ επικίνδυνες και θα έχουν ε, επιπτώσεις στο περιβάλλον των δύο χωρών, αλλά και στις κλιματικές αλλαγές. Και μάλιστα τώρα με την διάσκεψη για το κλίμα στο Ρίο θα πρέπει να πούμε τι ακριβώς κάνουμε για την εξισορρόπηση των μελλοντικών προοπτικών συνεργασίας σε ολόκληρο το, το γη. Και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κολομβία και το Περού. Επίσης θεωρούμε ότι μέσω της απελευθέρωσης της οικονομίας και έχουμε μιλήσει για αυτή την πτυχή στην τελευταία, στην 8η μάλλον υπουργική διάσκεψη στον ΠΟΕ, ότι χρειάζεται δηλαδή νέα προσέγγιση και θεωρώ ως εκ τούτου ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει λάβει υπόψη αρκετά την ε, τρέχουσα κρίση. Θεωρούμε επίσης ότι είναι ε, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το διαπραγματευτήκαμε με τους εκπροσώπους του παλαιού καθεστώτος και όχι με την σημερινή κυβέρνηση. Συνδέεται λοιπόν υπερβολικά με το παρελθόν και δεν εστιάζει αρκετά σε μελλοντικέ προοπτικέ. Τέλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, είχαμε διάφορες ευκαιρίες όπου έγιναν ανταλλαγέ απόψεων. Επίση πιστεύω ότι το ποτήρι είναι μισοάδιο και όχι μισογεμάτο. Και βεβαίως, ε, αν παραμένει οποιαδήποτε αμφιβολία στην Επιτροπή μας. ελπίζω πως με αυτό το ψήφισμα θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και να προετοιμάσουμε για την Επιτροπή και για την Ολομέλεια με τρόπο ώστε να έχουμε μια θετική προσέγγιση για αυτό το περίπλοκο θέμα. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο παρακαλώ. Uh, commission, uh, Η Επιτροπή. Ο κύριος Μικελάντζολο Μαργκερίτα. Thank um, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια για κάποια ζητήματα που ακούστηκαν συγκεκριμένα για τα βιοκαύσιμα όπως επίσης για τη φύση της ε, συνθήκης για τα προϊόντα βιοκαυσίμων. Θέλω να πω ότι η, συνθήκη, η, ε, συμφωνία συγγνώμη, από αυτή την έννοια είναι εντελώς ουδέτερη. Δηλαδή είναι μηδονικό ο για την είσοδο της αρνώσης βάση του GSP συν. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο τη Συμφωνία για τα ίδια τα βιοκαύσιμα, δεν υπάρχει καμία αλλαγή λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια που ακούστηκαν για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καταγράφουμε τα σχόλια που έγιναν η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει ο κόσμος ε, άρδιν τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά αυτές τις υπηρεσίε και να σα πω ότι στι συζητήσεις ε, που έλαβαν χώρα με το Περού και την Κολομβία είναι ε, συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει το 2007 και 2008. Άρα ελήφθη δεόντως υπόψη η παρούσα κατάσταση στι διαπραγματεύσει αυτές και βεβαίως ελήφθη υπόψη το συμφέρον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και του ευρωπαίου καταναλωτή. Ευχαριστώ. And, uh, Ο εισηγητής και πάλι για το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εντάχει, ευχαριστώ τον κύριο Λάγκα και τον κύριο Σούλτ και τους ε, σκιώδεις σε ό,τι αφορά την έκθεσή μου για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε, αν και κάποιες φορές ιδεολογικός πώς έχουμε διαφωνίες. Πάντως έχω την αίσθηση ότι κατανοούμε ο ένας τις ανησυχίες του άλλου. Αυτό που με ικανοποιεί περισσότερο είναι ότι όχι μόνο υπάρχει βούληση του Κοινοβουλίου να εστιάσει ιδίω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργατικών δικαιωμάτων, βιώσιμης ανάπτυξης κτλ. Αλλά ότι αυτό είναι μία ανησυχία που συμμερίζεται και η δημόσια διοίκηση και η κυβέρνηση για των δύο αυτών χωρών. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία στο να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το το αντικείμενο των συζητήσεων που θα έχουμε τον κύριο Λάγκα τις επόμενες τρεις ημέρες, ελπίζοντας την επόμενη φορά να έρθουμε εδώ με απαντήσεις. Όσο τρόπο να διασκεδάσουμε τις ε, ανησυχίες ε, ε, που ορθά έχουν κάποιοι συνάδελφοι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά ένα άλμα ποιοτικό σε αυτό το θέμα. Αλλά την άλλη να σε υπενθυμίσω και το εξής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει πίσω η συνθήκη ΙΠΑ Κολομβίας ε, τέθη σε ισχύ πριν από τρεις εβδομάδες και κάποια από τα ζητήματα που συζητούμε αυτή τη στιγμή είναι και προς όφελός μας, θα έλεγα, λόγω αυτή της θέσης ισχύ της ε, συμφωνίας με την ΕΠΑ. Δηλαδή πολλά από τα δικά μας αιτήματα ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε Κολομβία και Περού βάσει της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, γιατί έχουν κατανοήσει και οι δύο κυβερνήσεις ότι είναι υπέρ των λαών του. Πρόεδρε, μου επιβεβαιώνουν ότι η ψηφοφορία για αυτή την έκθεση θα γίνει στι 4.30 το απόγευμα, γιατί η Μερσή μιλάει για ενδεχομένη ψηφοφορία. Πρόεδρο, Η έκθεση δεν έχει ληφθεί υπόψη επισήμως από το Συμβούλιο. Έχει μόλις τώρα διαβιβαστεί. And uh, um, Και δεν έχει ακόμη μονογραφηθεί το κείμενο. Μπορούμε να ακολουθήσουμε την άγουσα σχετικά με την πολυτροπολογιών και σε αυτή την περίπτωση. Όχι. Όχι, θα το αφήσουμε, θα το αφήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση, γιατί ακόμη δεν έχει ε, λάβει γνώση επισήμως στο Συμβούλιο. Δεν Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε πρώτα ότι προβλέπει ο κανονισμός για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ποια είναι η πρόταση του εισηγητή που είναι θετική σε σχέση με αυτή την πρόταση. Ο εισηγητή και πάλι μου βεβαιώνει ότι αν ψηφίσουμε στις 4.30 το απόγευμα. Η απάντηση εκτό μικροφώνου. Uh, the uh, Mr. for item Ο κύριος Φιέλνερ για το σημείο 8 δεν είναι εδώ. Προχωρήσαμε πολύ γρήγορα σήμερα το πρωί. Ο ένας εκ των λόγο είναι προφανής. Φαίνεται ότι έχουμε αρχίσει ήδη τις διακοπές από πλευράς Ευρωβουλευτών. Θα διακόψουμε λοιπόν τη συνεδρίαση. Ολοκληρώνεται η συνεδρίαση για σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να προτείνω από τους συζητητές ε, εάν μπορούμε να κάνουμε λίγο νωρίτερα τη συνεδρίαση των συντονιστών για ένα τέταρτο μόνο, αντί για 11.30 να ξεκινήσουμε στις 11 και τέταρτο, Θα συζητήσω με τους υπόλοιπους συντονιστές για να γίνει νωρίτερα συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε το απόγευμα.